τους ή άλλους που να τους φροντίζουν. Αυτό είναι το πρόγραμμα που μας οδήγησε να προσκαλέσουμε σήμερα τους ε, διακεκριμένους προσκεκλημένους μας και να μας παρουσιάσουν τους κανόνες του, ε, του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου για να δούμε πώς οι κανόνες αυτοί μπορούν να επηρεάσουν το σημερινό μεταναστευτικό πλαίσιο. Χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις ήθελα να δώσω το λόγο στους πρώτους ομιλητές μας από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης και από το Πανεπιστήμιο των Βρυσαλίων. Έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ. Κυρίες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα επιφόρτησε με την εκπόνηση δύο εκθέσεων για τον τρόπο με τον οποίο οι κανόνε του ιδιωτικού δικαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, ώστε να αντιμετωπιστούν με συνεκτικότερο τρόπο τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό. Διαπιστώσαμε, μάλλον συγκροτήσαμε. Όχι, δεν είναι το σωστό PowerPoint, λυπούμε. Συγκροτήσαμε μία ομάδα από πανεπιστημιακούς, οι περισσότεροι είναι εδώ σήμερα. Το κατάλογο τον έχετε στο PowerPoint. Η πρώτη μελέτη έχει να κάνει γενικά με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ κανόνων διεθνούς ιδιωτικού δικαίου και των κανόνων σε σχέση με το δίκαιο για τους αλλοδαπούς και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά παιδιά μετανάστες ε, η δεύτερη μελέτη. Θέλουμε ε, να υπάρξει μεγαλύτερη αναγνώριση του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, προτείνουμε δράσεις για ευρωπαϊκό επίπεδο και έρευνες συμπληρωματικές που πρέπει να γίνουν. Τα ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσουμε είναι σημαντικά για να έχουμε ποιοτική μεταναστευτική πολιτική που θα ακτηρίζεται από συνέπεια και ανθρωπιά. Όμως, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίζουμε και είχαμε μόνο λίγε εβδομάδες για να πραγματευτούμε το θέμα. Καταλήξαμε σε διάφορα συμπεράσματα που ελπίζω ότι θα τα θεωρήσετε σημαντικά. Ουσιαστικά δεν μιλάμε για νομοθετικές, αναλυτικές νομοθετικές προτάσεις, γιατί γι' αυτό πρέπει να γίνουν συμπληρωματικέ έρευνε. χρησιμοποιήσαμε την ομολογία καθώς ε, και τη θεωρία και τη συμπληρώσαμε με συνεντεύξεις από τα διάφορα κράτη-μέλη, με τον Ερυθρό Σταυρό, τις υπηρεσίες παιδικής μέρημνας, ε, κεντρικές αρχές, ε, καθώς επίσης και με τις αρμόδιες αρχές για θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Οι συνεντεύξεις αυτές έδειξαν ότι δεν υπάρχει συντονισμός των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και του δικαίου περί αλλοδαπών, αλλά ότι υπάρχει δυνατότητα να τον έχουμε αυτόν τον συντονισμό. Και αυτό θέλουμε να το καταδείξουμε με τις δύο μελέτες. Θα δώσω όμως το λόγο στη συνάδελφό μου τώρα, για να σας πω τα υπόλοιπα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, θέλω να σας παρουσιάσω συντομία τη μελέτη για το διωτικό διεθνέ δίκαιο στο πλαίσιο της αυξανόμενη κινητικότητα με στόχο να σας πούμε ποιε είναι οι αλληλεπίδράσει μεταξύ μεταναστευτικού δικαίου και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που διέπει ε, άτομα τα οποία έρχονται από τρίτες χώρες και το μεταναστευτικό ρυθμίζει τι γίνεται μεταξύ των κρατών μελών της ζωή, δηλαδή ε, μεταξύ κρατών μελών. Όλα αυτά εντάσσονται στο χώρο ελευθερίας ασφάλειας δικαιοσύνης. Είδαμε ότι δεν υπάρχει όμως μια κοινή προσέγγιση και κάθε τομέα έχει τους δικούς του κανόνες. Έχουμε τους μετανες και του κανόνε περί ε, αστικής προστασίας ή του κανόνε διεθνού ιδιωτικού δικαίου που πολλέ φορέ είναι τελείω διαφορετικοί. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι μια καλύτερη αλληλεπίδραση αυτών των δύο τομέων είναι ευκταίο, κάτι ευκταίο που δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε άλλο. Θα έρθω και σε κάποια βασικά πορίσματα της μελέτης, αλλά καταρχάς θέλω να σας πω ότι η μελέτη αυτή δεν είναι παρά μία πρώτη διερευνητική προσπάθεια και χρειάζεται σε βάθος έρευνα, συμπληρωματική έρευνα. Θα ήταν πολύτιμο κάτι τέτοιο. Η μελέτη λοιπόν έχει τρία κεφάλαια. Το πρώτο είναι αναγνώριση το καθεστώτος των προσώπων, το δεύτερο είναι η εφαρμογή του Διεθνού και το τρίτο έχει να κάνει με τη σύμβαση για του πρόσφυγε τη ε, Σύμβαση τη Γενέβη. Ελπίζουμε ότι θα μα στηρίξετε να βρούμε λύσει που θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την αναποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο δεσμών κανόν, δηλαδή διεθνέ ε, ιδιωτικό δίκαιο από τη μία και μεταναστευτικό από την άλλη. Γιατί παραλαμβάνω ότι με την λεπίδραση και το σεβασμό τη προσωπική και κοινωνική ζωή, θα φέρουμε τα καλά αποτελέσματα. Πριν έρθω στα βασικά απορίσματα όμω, να ξεκινήσω με κάποιε ερωτήσει που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα, με την πραγματική ζωή και δείχνουν πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα και πόσο μεγάλε είναι οι προκλήσει που αντιμετωπίζει το Διεθνέ Ιδιωτικό Δίκαιο σε αυτό το πλαίσιο τη μετανάστευση. Ένα παράδειγμα. Ένα σωμαλό αγόρι. Πώ αν δεν έχει πιστοποιητικό γέννηση μπορεί να αποδείξει ότι ανήκει σε μια μειονότητα, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να έχει έναν κηδεμόνα. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε χώρες που δεν υπάρχουν ληξιαρχικές υπηρεσίες συστηματικές. Άρα, Γενάρη ή Ιούνιο φαίνεται να έχουν γεννηθεί όλα τα παιδιά, διότι δεν υπάρχει, μόνο τότε γίνονται οι καταγραφές ληξιαρχικές. Και δεν ξέρουμε λοιπόν αν ένα άτομο είναι ε, σε μια άνοιξη μειονότητα και χρειάζεται ε, επιμέλεια κάποιον κηδεμόνα που θα τον εκπροσωπήσει στις διαδικασίες για την παροχή ασύλου για παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα είναι, έχουμε ένα Αφγανό ζευγάρι που ζητά άσυλο και δίνει ένα πιστοποιητικό γάμου που λέει ότι έγινε συσκευτικός γάμος όταν όμως το κορίτσι ήταν 16 και, παρακα... και λίγο. Πώς ε, όμως μπορούμε να ε, αποδείξουμε κάτι τέτοιο ή παραδείγματο χάρη ένα κορίτσι που γεννήθηκε μέσα στα, στους καταβλισμούς ε, ε πώς μπορεί να αποδείξει ότι αυτό το παιδί, παραδείγματος ε, ο πατέρας του ανήκει αυτή τη στιγμή που δεν έχει πιστοποιητικό ή ένα κορίτσι από το Κονκό που το θετεί της στη Γαλλία και δεν του δίνουν θεώρηση για να πει στη Γαλλία κτλ. κτλ. Πώς λοιπόν αξιολογούνται τα αλλουδαπά έγγραφα που έχουν να κάνουν με την κατάσταση την οικογενειακή ε, κάποιο άτομο. Ένα έγγραφο από τη Συρία, όπως αυτά που βλέπετε, ή ένα πιστοποιητικό γάμο όπω αυτό που βλέπετε τώρα από το Αφγανιστάν. Πώ μπορεί κανεί να τα διαβάσει πόσο δεν υπάρχουν δε ε, έγγραφα και επικυρωμένα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιε ε, για θέματα αστικού δικαίου και μεταξύ των μεταναστευτικών αρχών και των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνε για τα ζητήματα ε, αστικού δικαίου. Εννοούμε ληξιαρχικέ αρχέ, αρχέ παιδική προστασία κτλ, κτλ. Αυτά είναι τα βασικά πορίσματα του κεφαλαίου 1 Εκεί αναλύεται αυτό το ε, θέμα της αναγνώρισης ε, του προσωπικού, της προσωπικής κατάστασης ε, που, που αποκτάται στο εξωτερικό. Και βλέπουμε εδώ κάποιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο τομέων που προανέφερα, οικογενειακή επανένωση, προστασία των ασυνόδευτων παιδιών, που πρέπει όμως να αποδείξει κανείς ότι ανοίξει μια μειονότητα, πρέπει να έχει ένα πιστοποιητικό γέννηση. Αλλά έχουμε δύο διαφορετικέ δέσμε κανόνων που, όπω είπαμε, ναι, να αλληλεπιδρούν, μπορεί λοιπόν, να έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα. Σε κάποιε περιπτώσει, η αναγνώριση ε, με βάση τους κανόνες του Διεθνού Συντηρητικού Δικαίου είναι προϋπόθεση για να πάρει κανεί το καθεστώς ε, του μετανάστη σε μια χώρα. Ενώ σε άλλε περιπτώσει δεν υπάρχει Καθεστώ μετανάστη. Παρά την αναγνώριση του καθεστώτος κάποιου, της κατάστασης κάποιου δυνάμει του, διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Παραδείγματο χάρη η υιοθεσία στην Αλλοδαπή, αλλά όχι η άδεια παραμονή για το παιδί. Για να δείτε πόσο πολύπλοκο είναι το θέμα που συζητάμε. Ε, και για να σα δώσω κι άλλο ένα παράδειγμα για την αναγνώριση της προσωπική κατάστασης ε, δυνάμει του Διεθνού Ιδιωτικού Δικαίου. Ω προπόθεση για την αποκτήση του καθεστώτο του μετανάστη. Θέλω να σα μιλήσω για κάποιε μεταφορές δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου που γίνονται μόνο αφού έχει υπάρξει αναγνώριση ενό ξένου πιστοποιητικού γάμου γέννηση. Η γενική επανένωση είναι εφικτή μόνο αν υπάρξει αναγνώριση ενό ξένου πιστοποιητικού γάμου. Στην πράξη υπάρχουν μείζωνα προβλήματα. Λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία αποδεικτικά για τους οικογενειακούς γονικούς δεσμούς, για το γάμο κτλ. κτλ. Και στη μελέτη μας ε, προτείνουμε εναλλακτικέ μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούνται επί του παρόντος όταν λείπουν ε, σημαντικά προσωπικά έγγραφα. Βρήκαμε λοιπόν καλές πρακτικές σε κάποια κρατημέλη, όπως για παράδειγμα στη Γαλλία, η Όφπρα έχει κάποια έγγραφα για τα άτομα που παίρνουν διεθνή προστασία όταν δεν έχουν έγγραφα που να αποδεικνύουν την προσωπική του κατάσταση. Καλέ οι πρακτικέ αυτέ μεν, όμω μεγάλε οι διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών δε. Ή υπάρχουν περιοριστικέ πρακτικέ που δείχνει ότι υπάρχει καχυποψία απέναντι στι υπηκόστρε των κρατών, ότι δόχο έχουν να εξαπατήσουν τι αρχέ. Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων που θα αντικαταστήσουν τα χαμένα έγγραφα. Κατάλληλες όμως, επαρκείς εναλλακτικές μεθόδους ε, με διαδικαστικές εγγυήσεις που θα είναι ομοιόμορφες επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι για σας, ε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές. Μια, ένα βασικό πόρισμα της μελέτης αυτής αλλά και της έκθεσης ε, που θα παρουσιάσει στην άρθρο Σαμπίν έχει να κάνει με την ε, πολιτισμό της ηλικία ε, και το αν ανήκει κάποιος σε μια μειονότητα. Αν θεωρείται αναξόπιστο, το πιστοποιητικό αν δεν υπάρχει πιστοποιητικό γέννησης. Και πάλι εδώ αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Προσπάθειε για να υπάρξει μεγαλύτερη ομοιομορφία τη διαδικασία πολιτισμού τη ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι κατεπήγον οι διαδικασίε πολιτισμού τη ηλικία θα πρέπει βέβαια να σέβονται τα συμφέροντα του παιδιού σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Και τα αποτελέσματα τέτοια διαδικασία θα πρέπει να είναι αποδεκτά σε όλα τα κράτη-μέλη, από όλε τι αρχέ. Και έρχομαι τώρα στο δεύτερο, που είναι αναγνώριση του προσωπικής κατάστασης, πάλι ε, δυνάμει του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου, που δεν αρκεί όμως από πλευράς μεταναστευτικού δικαίου. Δηλαδή, ναι, μην υπάρχει αναγνώριση, αλλά δεν δίνεται το καθεστώ του μετανάστη. Θα δείτε και στη μελέτη μας ότι είναι αναποτελεσματική αλληλεπίδραση των δύο αυτών. Δηλαδή, μεταναστευτική μεταναστευτικής και διεθνού ιδιωτικού δικαίου. Θα σας μιλήσω για έναν Ισλαμικό οργανισμό που δείχνει πόσο δεν υπάρχει ε, συντονισμός μεταξύ των δύο δεσμών ε, κανόνων. συστηματικά δεν υπάρχει δυνατότητα για το παιδί να εισέλθει και να διαμένει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχομαι στο έβδομο βασικό πόρισμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εν... να εφαρμόσει την Σύμβαση του 1996 της Χάγης και τις υποχρεώσεις που επιβάλλει στα κράτη-μέλη στην περίπτωση ανηλίκων, π.χ. στην περίπτωση της Κάφαλα. Κάφαλα παρά το ότι δεν υπάρχει στο δίκαιο των ευρωπαϊκών κρατών δημιουργεί κάποια δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε δηλαδή ότι τα παιδιά θα πρέπει να λάβουν βίζα ή άδεια παραμονή, αν είναι να γίνει σεβαστό το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Τέλος, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το δεύτερο κεφάλαιο σε αυτή τη μελέτη για την εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου. Στο πλαίσιο τη μετανάστευση υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες για την εφαρμογή του αλλοδαπού δικαίου. Ιδιαίτερα από την σκοπιά των μη δικαστικών αρχών, όπως ε, από τον ληξίαρχο, ή από τις αρχές της αρμόδιας για τη μετανάστευση. Παραδείγματος χάρη, όταν έρχεται ένας μετανάστης στα σύνορα, ο συνοριοφύλακας ε, ίσως πρέπει να αξιολογήσει την αυθεντικότητα ε, εγγράφων ταυτότητας σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης ίσως πρέπει να αποφασίσουν ε, οι αρχές για γάμους οι οποίοι θα είναι θρησκευτικοί ή γάμοι με παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. και βεβαίως θα πρέπει να κρίνουν οι αρχές που εφαρμόζουν τον κανονισμό του Δουβλίνου το εάν απαιτείται η εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου για την περίπτωση γάμου ή άλλων ληξιαρχικών πράξεων. Εδώ πέρα λοιπόν γύρονται κάποια φλέγοντα ζητήματα. Οι αρχές έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν το αλλοδαπό και αν ναι πώς ή γνωρίζουν καν το ζήτημα αυτό διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχει κάποια επιστημονική έρευνα για αυτά τα φλέγοντα ζητήματα. Η μελέτη αυτή παρέχει μόνο την εικόνα κάποιων κρατών μελών. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην συνάδελφό μου. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η δεύτερη μελέτη επίσης αφορά την αλληλεπίδραση του μεταναστευτικού δικαίου και του ιδιωτικού διεθνούς εστιάζοντας ειδικότερα στην προστασία των παιδιών. Συγκεκριμένα ασχολείται με την προστασία ε, ή ανηλίκων οι οποίοι μετακινούνται χωρίς κάποιον ε, κηδεμόνα. Το πεδίο εφαρμογής ε, της μελέτης είναι ευρύτατο γιατί αφορά όλα τα συνόδευτα ανήλικα είτε ζητάνε άσυλο είτε όχι ανεξαρτήτως δηλαδή του εάν φεύγουν από διώξεις ή όχι. Η οχι Μία αφετηρια της μελέτης μας είναι το ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ε, δύο ε, αυτών πεδίων της νομοθεσίας του μεταναστευτικού δικαίου και του διεθνούς ε, ιδιωτικού δικαίου. Αλλά υπάρχουν κανόνες για την προστασία των ανηλίκων και στις δύο περιπτώσεις, αλλά με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι οι κανόνες αυτοί λειτουργούν ε, σε τελείως διαφορετικά σύμπαντα. Δεν είναι συντονισμένοι και αγνοούν τελείως το ένα το άλλο. Αυτό βεβαίως είναι ενισχυτικό και άρα τα βασικά ευρήματα της ε, μελέτες μας αφορούν ακριβώς το πώς θα υπάρχει κάποιος συντονισμός. Ευτυχώς υπάρχει ο κανονισμός Βρυξελών 2 για τις υποχρεώσεις ε, των γονέων και το μέσο του κοινού συστήματος ασύλου, τα οποία αναθεωρούνται αυτή τη στιγμή, οπότε υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή να βελτιωθεί η κατάσταση. Η μελέτη μας, λοιπόν, χωρίζεται σε ε, τρία κεφάλαια. Το ένα αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ διεθνούς ιδιωτικού και μεταναστευτικού δικαίου, το άλλο αφορά τους διασυνοριακούς μηχανισμούς ε, συνεργασίας και το άλλο αφορά τα οριζόντια ζητήματα που αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Θα περιοριστώ λοιπόν στα πιο σημαντικά ευρήματα στα κεφάλαια 1 και 2. Πρώτα απ' όλα, για την αλληλεπίδραση διεθνούς ιδιωτικού και μεταναστευτικού δικαίου. Θα ήθελα να τονίσω το, ε, το έβριμα υπαριθμών 3. Ζητάμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ του κανονισμού Βρυξελών 2α και του μέσου του κοινού Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ασύλου. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα συνόδευτο παιδί από το Ιράκ που ζητάει άσυλο. Θα πρέπει να του οριστεί κίδεμόνας που θα το εκπροσωπεί στην διαδικασία και αυτή τη στιγμή έχει κάθεστος πρόσφυγα πρέπει να υπάρξει μια μακροπρόθεσμη λύση. Αν αντιθέτω δεν λάβει το καθεστώς πρόσφυγα, επίσης πρέπει να βρεθεί μια λύση μόνιμη ε, προς τα συμφέροντα του παιδιού. Ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο. Ποιο κράτος μέλος έχει την δικαιοδοσία να λάβει τέτοια μέτρα προστασίας. Ο κανονισμός του Δοβλίνου προβλέπει κανόνες που ισχύουν στην διαδικασία ασύλου, ενώ ο κανονισμός Βρυξέλλες 2α ε, περιέχει τους γενικούς κανόνες για την προστασία παιδιών ε, σύμφωνα με το αστικό δίκαιο οι οποίοι ισχύουν υπό οποιασδήποτε συνθήκε και για παιδιά που ζητούν άσυλο. Όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, οι συγκεκριμένες ε, διατάξεις για το άσυλο φαίνεται ότι κατησχύουν του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου. Τουλάχιστον όσο εκκρεμεί η αίτηση ασύλου. Όμως η κατάσταση δεν είναι απολύτως σαφής και η προστασία των ανηλίκων δεν είναι η βέλτιστη. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι οι διασταυρώσεις θα πρέπει να γίνουν στον κανονισμό Βρυξελών 2α και στο μέσο CAS για να καθοριστούν οι αλληλεπιδράσεις. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού Βρυξελών 2α θα πρέπει να δώσουμε βάρος στις ιδιαίτερες ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων. Και αυτό βεβαίως απαιτεί συντονισμό με τους κανόνες που υπάρχουν ήδη στο πλαίσιο του κοινού συστήματος ασύλου. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της ε, αναθεώρησης του κοινού συστήματος ασύλου πρέπει να δοθεί βάρος ε, στα μέσα που υπάρχουν ήδη στο πλαίσιο του αστικού δικαίου, δηλαδή τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α, αλλά και σε σχέση με τα τρίτα κράτη, τη σύμβαση της Χάγης του 1996 για την προστασία ανηλίκων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ε, τωρινής κρίσης, πρέπει να μην παραβλέπουμε την ανάγκη για προστασία των ανηλίκων που δεν ζητούν άσυλο. Ας ε, δούμε το παράδειγμα τον κανόνα περί δικαιοδοσίας του άρθρου 13 του κανονισμού των Βρυξελών 2α, που έχει μεγάλη σημασία για τους ασυνοδευτούς ανήλικους. Αφορά ακριβώς ε, την ε, παρουσία του παιδιού. Η παράγραφος 2 είναι ένα από τα λίγα παραδείγματα όπου το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο αναφέρεται συγκεκριμένα στην κατάσταση ανηλίκων μεταναστών. Τι γίνεται όμως ε, για την περίπτωση ατόμων που μεταναστεύουν για λόγους οικονομικούς και όχι για λόγους δίωξης. Ας ε, φανταστούμε έναν ασυνόδευτο ανήλικο όχι από το Ιράκ αλλά από το Μαρόκο Μπορεί αυτό το παιδί να θεωρηθεί εκτοπισμένο λόγω προβλημάτων στη χώρα του. Εγείρεται αυτό το θέμα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Βρυξέλλες 2α αλλά και τη Σύμβαση της Χάγης του 96 γιατί υπάρχουν και εκεί παρόμοιες διατάξεις. Στη μελέτη μας προτείνουμε το άρθρο 13 και η ανάλογη διάταξη της ε, συνθήκης της Χάγης ε, να ερμηνεύονται με τρόπο ο οποίος θα είναι πιο ελαστικός, δηλαδή ανεξαρτήτως για τον λόγο για τον οποίο έχει μετακινηθεί ο ανήλικος. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το κείμενο δεν είναι σαφές. Η συγκεκριμένη ε, κατάσταση του κάθε παιδιού απαιτεί περαιτέρω προσοχή. Το δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης μας αφορά την διασυνοριακή συνεργασία και τους σχετικούς μηχανισμούς που έχουν σημασία για την αποτελεσματική προστασία των παιδιών αυτών. Ε, σημασία λοιπόν έχει συνεργασία για να βρεθούν πληροφορίες για την κατάσταση του ανηλίκου και της οικογένειάς του. Για να επανέλθω στο παράδειγμα ενός ανηλίκου από το Ιράκ που βρίσκεται παραδείγματος χάρη σε ένα κέντρο υποδοχής στην Ελλάδα απαιτείται να εντοπιστούν οι γονεί του και άλλοι συγγενείς μπορεί να είναι δυσπαρμένοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης απαιτείται συνεργασία όταν οι αρχές ε, εξετάζουν την μεταφορά του παιδιού σε άλλη χώρα που μπορεί να είναι η χώρα προέλευσης ή ένα κράτος μέλος ή ένα τρίτο κράτος όπου βρίσκονται μέλη της οικογένειας του ανηλίκου. Παραδείγματος χάριν, τα παιδιά του εν λόγω Ιρακινού μπορεί να βρίσκονται ακόμα στο Ιράκ και βεβαίως δεν τίθεται ζήτημα επιστροφής στην χώρα προέλευσης, αλλά ένας αδερφός του μπορεί να ζει παραδείγματος χάρη σε άλλο κράτος μέλος και ίσως είναι προς το συμφέρον του παιδιού να μην παραμείνει στην Ελλάδα ασυνόδευτος, αλλά να πάει με τους συγγενείς του σε άλλη χώρα. Θα ήθελα εδώ να τονίσω το τέταρτο πόρισμά μας πρόταση της Επιτροπής για την αναδιατύπωση του κανονισμού των Βρυξελών 2α. Το κεφάλαιο για τη συνεργασία μεταξύ κεντρικών αρχών και διοικητικών αρχών δεν είναι αποτελεσματικός, οπότε ο μηχανισμός δεν έχει λειτουργήσει στο πλήρες δυναμικό του. Η πρόταση της Επιτροπής εντοπίζει περιοχές συνεργασίας που θα επιτρέψουν να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών. Οπότε πρέπει να υπάρξει σοβαρή στήριξη. Πάντω, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο κανονισμό Βρυξελών 2 ε, ισχύει για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ενώ η προστασία των παιδιών μεταναστών έχει περισσότερο να κάνει με συνεργασία με τρίτα κράτη, με αρχέ τρίτων κρατών, ε, κράτη προέλευση, κράτη διέλευση κτλ. Η συνεργασία με τα τρίτα κράτη διεπεται από την Σύμβαση του 1996 της Χάγης για την προστασία των παιδιών που είναι εφαρμοστέα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κυρωθεί από άλλα 18 κράτη μεταξύ των οποίων η Τουρκία, η Αλβανία και το Μαρόκο. Ως προς την Σύμβαση της Χάγης θα ήθελα να αναφέρω το τρίτο πόρισμά μας η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει καταρχάς να βεβαιωθεί ότι τα κρήτα κράτη που ήδη είναι συμβαλόμενα μέρη στην ε, σύμβαση την εφαρμόζουν ορθώς. Εφόσον αυτό δεν συμβαίνει, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει συνδρομή στα κράτη αυτά. Διότι η κύρωση της σύμβασης δεν αρκεί από μόνη της ως κίνηση. Δεν σημαίνει ότι ε, ε, ισοδυναμεί με πλήρη εφαρμογή. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντοπίσει εκείνα τα κράτη-μέλη, εκείνα μάλλον τα τρίτα κράτη, με τα οποία απαιτείται συνεργασία για την προστασία των ασυνόδευτων αελίκων ή δυνατών και να τα ενθαρρύνει να συμπληθούν στην Σύμβαση του 1996. Για να ολοκληρώσω. Για να ολοκληρώσω, θέλω να τονίσω ότι στην έρευνά μας βρήκαμε πολλά ενδιαφέροντα εργαλεία τα οποία είτε ήδη έχουν προβλεφθεί, είτε συζητώνται στα πλαίσια της διαδικασίας του ΡΙΚΑ, της αναδιατύπωσης. Εδώ και το δίκαιο περί μετανάστευσης και το διεθνές ιδιωτικό μπορούν να χρησιμεύσουν, αλλά είναι σε τελείως ε, διαφορετικές και αποκλεισμένες μεταξύ τους σφαίρες. Δεν συνδυάζονται, πράγμα που θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο. Γι' αυτό χρειάζεται εδώ η παρέμβαση του Ευρωπαίου Νομοθέτη και γι' αυτό το σκοπό εντοπίσαμε στις δυο μας μελέτες συγκεκριμένα σημεία δράσης Βεβαίω, είμαστε δεσμευμένοι να συνεχίσουμε την έρευνα σε αυτόν τον κλάδο, διότι πιστεύουμε ότι πολλά μπορούν να γίνουν ακόμη για να πετύχουμε καλύτερη διασύνδεση των δύο νομικών πλαισίων με καλύτερα αποτελέσματα. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ σας. Ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ. Τώρα θα, θα συνεχίσουμε το δεύτερο μέρο του εργαστηρίου μα. με τη Μαρτίνα Χέρμπ Κλούνεμαν, δικαστή και μέλο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, η οποία θα μα μιλήσει για την εμπειρία τη στον χώρο αυτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που, που μου ζητήσατε να συντάξω μία έκθεση ε, ως ε, μία δικαστής ε, σε δικαστήριο που δικάζει οικογενειακές υποθέσεις. Ασχολούμαι με την πράξη, στην πράξη με αυτά τα ζητήματα κάθε μέρα με ανηλίκους, με αλλοδαπούς, με αλλοδαπούς ανηλίκους. Έχω λοιπόν όλες αυτές τις εμπειρίες ε, που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας από τις αποφάσεις ε, των δικαστηρίων που είναι δημόσιες. Ε, μου έχουν απευθύνει πάρα πολλά ερωτήματα και Ευρωπαίοι δικαστές καθώς είμαι σύνδεσμος και στο Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και στο Δίκτυο της Χάγης και βεβαίως είμαι μία από τις λίγες δικαστές που στην αρχή έλεγε ότι κάτι έπρεπε να γίνει και ότι υπήρχε κάποιο αντικείμενο εδώ πέρα. Λοιπόν, στη Γερμανία η προσέγγιση είναι η εξής στο δημόσιο δίκαιο. Προέχει η προστασία του ανηλίκου. Δηλαδή όταν έχουμε έναν ασυνόδευτο ανήλικο ε, πρόσφυγα ενώπιόν μας ε, Έχουμε πρώτα απ' όλα το ότι έχουμε μπροστά μας μια ανθρώπινη ζωή, ένα παιδί, έναν ανήλικο, το οποίο, ο οποίος δεν έχει ικανότητα δικαιοπραξίας, άρα απαιτείται ένας κηδεμόνας και μια προστασία. Και μετά έρχεται ε, σε δεύτερη μοίρα το ότι πρόκειται περί αλλοδαπό και άρα ισχύει το δίκαιο περί αλλοδαπών. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τη νέα παράγραφο στον ε, κώδικα περί κοινωνικής ασφάλισης ε, που εισήχθη το 2015 όταν ήρθαν πολλοί πρόσφυγες. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα εντός της Γερμανίας ε, που αφορά ακριβώς την αναδοχή αυτών των παιδιών και έχουμε δύο υπηρεσίες που ενημερώνουν πρώτα απ' όλα την λεγόμενη υπηρεσία ανηλίκων και μετά υπάρχει μια κλίδα κατανομής ε, σύμφωνα με την οποία η υπηρεσία ανηλίκων βάζει τα παιδιά αυτά σε ανεδοχές οικογένειες. Με το νέο σύστημα έχουμε αυτό το οποίο ε, ρυθμίζει ο νόμος, ε, δηλαδή το να οριστούν πρώτα απ' όλα οι υπηρεσίες ανηλίκων ως κηδεμόνες και εκπρόσωποι του παιδιού. Δηλαδή η υπηρεσία ανηλίκων μετά κατά κανόνα πρέπει να ενημερώσει το δικαστήριο ανηλίκων το οποίο ορίζει τον ορισμό ενός κηδεμόνα. Το γερμανικό οικογενειακό δίκαιο δεν άλλαξε στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης, δεν υπήρχε ανάγκη για κάτι τέτοιο. αν υπάρχει ανάγκη προστασίας ενός ανηλίκου δεν παίζει κάποιο ρόλο η υπηκότητά του. Ο καθένας μπορεί να το γνωστοποιήσει στις αρχές. Κατά κανόνα βεβαίως πρόκειται για την υπηρεσία ανηλίκων όπως είπαμε, αλλά μπορεί να είναι πιθανόν να μας ειδοποιήσουν ε, συγγενείς για κάποιες περιπτώσεις. Εφόσον λοιπόν μιλάμε για ανηλίκους, οι οποίοι έχουν περιορισμένη ικανότητα δικαιοκρατία, Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να οριστεί σε ασυνόδευτο ανήλικο κάποιος ε, εκπρόσωπός του, ένας κηδεμόνας ο οποίος ε, θα μπορεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του παιδιού. Εάν δεν υπάρχει κηδεμόνας, τότε ορίζει κάποιον ε, ε, η αρμόδια αρχή το δικαστήριο. Η ιδιαιτερότητα στο γερμανικό σύστημα είναι η εξής. ότι όταν ερχόμαστε εμείς ε, σε επαφή με τα παιδιά ε, τότε αυτοί οι ενήλικοι βρίσκονται λίγες εβδομάδες ή λίγους μήνες στην Γερμανία. Δηλαδή βρίσκονται στη Γερμανία αλλά είχαν μέχρι τότε συνήθι τόπο κατοικία στην, χώρο, στην χώρα προέλευσης τους. Οπότε τότε εφαρμόζουμε το άρθρο 13 παράγραφο δύο, αλλά η ιδιότητα του πρόσφυγα δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δικαιολογήσει την παραναμονή του στην ε, χώρα. Αν βρίσκεται πούμε, για περισσότερο καιρό μπορεί να ισχύσει το άρθρο 8 του κανονισμού των Βρυξελών. Στην πράξη είναι δύσκολο να καθορίσουμε ποιος είναι πρόσφυγας ποιος έχει φύγει λόγω ταραχών ή ποιος απλά έφυγε από το σπίτι του. Δεν έχουμε δυνατότητες να εξετάσουμε κάτι και ουσιαστικά εξαρτώμεθα από τα όσα μας λέει ο ίδιος ο ανήλικος. Το γερμανικό δίκαιο λέει ότι όταν το δικαστήριο διαπιστώνει ότι οι γονείς δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, την επιμέλεια δηλαδή του παιδιού, τότε θα πρέπει να ορίσει το δικαστήριο κάποιον και δαιμόνα. Αυτή είναι η νομική βάση. Υπάρχουν βεβαίως κάποια προβλήματα που προκύπτουν στην πράξη και τα έχω τονίσει και προσπάθησα να σας παρουσιάσω το τι θεωρώ εγώ λογικότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι, λογικοί, όλοι οι Γερμανοί δικαστέ ακολουθούν την δική μου λογική και καμιά φορά υπάρχει η αβεβαιότητα. Λοιπόν, έχουμε πρώτα απ' όλα την διαπίστωση τη ηλικία. Κατά κανόνα δεν υπάρχουν έγγραφα. Ίσως να υπάρχει στο κινητό μία φωτογραφία ενός εγγράφου και ακόμα και αυτό δεν ξέρουμε αν είναι γνήσιο. Τι κάνουμε τότε. Πρέπει εμείς να ερευνήσουμε και Βεβαίω, ε, πάντα προς ε, όφελος ε, του ετούμενου. Αλλά βέβαια υπάρχει και κάποιο όριο, πιο καθορίζουμε το όριο. Επίσης, πού βρίσκουμε αυτές τις πληροφορίε, ή μπορεί να υπάρχουν, παραδείγματο χάρη, αποφάσει αλλοδαπών δικαστηρίων. Επίσης, πώς διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούν να ασκήσουν οι γονεί την επιμέλεια. Συχνά, ανήλικοι μας λένε ότι έχουν επαφές μέσω κινητού ή υπολογιστή με τους ε, δικούς τους ε, καμιά φορά και κάθε μέρα. Μπορεί έτσι να ασκήσουν επιμέλεια. Άλλοι έρχονται στην Ευρώπη και έχουν μια, μια γραπτή εξουσιοδότηση. Είτε μιλάμε για άτομα που τους συνοδεύουν ή ιδιαίτερα για άτομα τα οποία βρίσκονται ήδη στην Ευρώπη και εκεί πέρα θέλουν να πάνε τα παιδιά. Επαρκεί κάτι τέτοιο. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Βεβαίως... Ε, πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε το ποιος ε, θα είναι ο Επίτροπο ο οποίος ε, θα αναλάβει το παιδί. Βεβαίω το θέμα δεν αφορά μόνο την οικογενειακή επανένωση. Υπάρχουν ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη το αναλάβει ο ανήλικος ε, οικονομική στήριξη ή αν πρέπει να εγχειριστεί. Θα πρέπει να γραφτεί στο σχολείο, πρέπει να μάθει μια τέχνη. Και μετά τελείως ε, ατομικά ζητήματα ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Ποιες είναι οι απαιτήσει λοιπόν για κάποιον ε, κίδεμονα. Ε, δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολα ε, να πληρεί κάποιος όλες αυτές τις απαιτήσει. Δηλαδή να έχει παιδαγωγικές γνώσεις, πολιτισμικές γνώσεις, να γνωρίζει το δίκαιο περί αλλοδαπών, την κινδύνους περί τράφικινγκ, γλώσσες τουλάχιστον αγγλικά που θα μιλάνε οι ανήλικοι κατά κανόνα. Καλό θα ήταν βεβαίως να είναι κάποιος ο οποίος μιλάει και τη μητρική γλώσσα του ανηλίκου. Δύσκολο είναι βεβαίως και το πότε ενηλικιώνεται ο ανήλικος. Συγγνώμη, δεν δουλεύει το... Λοιπόν, το ερώτημα είναι... Να το. Ισχύει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το γερμανικό δίκαιο, το διεθνές ιδιωτικό ή το δίκαιο της χώρας προέλευσης, γιατί σε άλλες χώρες δεν είναι 18 η ενηλικίωση ή η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Περιπροσφύγων. Λοιπόν, οι διάφορες ε, δυνατότητες ε, για άδεια παραμονή στη Γερμανία αναφέρθηκαν ήδη. Σύντομα. Το 2015 στην κορύφωση του μεταναστευτικού κύματος ε, η ικανότητα δικαιοπραξίας των ανηλίκων ανέβηκε από τα 16 στα 18 ακριβώς για να δοθεί προβάδισμα στην προστασία των ανηλίκων. Οπότε, συνολικά έχουμε μια διτή προσέγγιση. Έχουμε το ε, δημόσιο και αστικό και ποινικό δίκαιο. Κάτι πολύ επίκαιρο, 2 Ιουνίου 2017 η Γερμανική Βουλή ενέκρινε τον νόμο απαγόρευσης γάμου ανηλίκων. Και θα σας πω πως έχει. Κατά την άποψή μου, ο τρόπος αντιμετώπισης ε, ανηλίκων ε, σέβεται τα δικαιώματα των ανηλίκων. Οι αλλαγές ε, του νόμου έχουν εξεταστεί από επιστημονικές επιτροπές, αλλά βεβαίως πρέπει να απαντηθούν πολλά ανοιχτά ζητήματα και να βελτιωθεί η κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Όλες οι παρεμβάσεις ήταν ε, πολύ σημαντικές και διαφωτιστικές, κυρίως υπό το φως της ε, τωρινής της παρούσας περίοδου που είναι ιστορική, γιατί προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μεταναστευτικές ροές και η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Ιδίω με τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος για το Άσυλο. Είναι πολύ ε, χρήσιμη πρόταση να συμπεριλάβουμε τις δισταυρούμενες αυτές αναφορές ε, στις Βρυξέλλες 2 και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Θα τις σκεφτούμε σοβαρά αυτές τις προτάσεις σας και επί ευκαιρία της μεταρρύθμισης ε, που βρίσκεται υπό συζήτηση αυτή τη στιγμή. Οι προεκτάσεις και οι αλληλοσυσχετισμοί είναι προφανείς. Τα αναφέρατε κι εσείς Πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να εντοπιστεί η ακριβής ηλικία του ανηλίκου. Σε ένα λόγου χάρη πιστοποιητικό γάμου. Προβλήματα τα οποία τα κράτη-μέλη τα αντιμετωπίζουν πλέον καθημερινά και τα οποία επιφέρουν επιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο. Όχι μόνο στις σχέσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και των εξωευρωπαϊκών με τις ευρωπαϊκές. Σε ό,τι αφορά την guardianship, την επιμέλεια των ασυνόδευτων ανηλίκων, είναι ακόμη πιο ευαίσθητο το θέμα. Ακόμη πιο ευαίσθητο, διότι σήμερα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που φτάνουν στην Ευρώπη, ή μάλλον ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που φτάνει στην Ευρώπη, αυξάνεται διαρκώς και δυστυχώς Δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ε, επιτρόπων ή κυβεμόνων ή υπευθύνων που θα φροντίσουν αυτούς τους ασυνόδευτους ανήλικους που έρνουν και σε μεγάλους αριθμούς. Η περίπτωση όμως των ασυνοδευτών ε, ανηλίκων θα πρέπει κάπως να ληφθεί υπόψη και ίσως ε, εθελοντικά ή οικειοθελώς να αναλαμβάνεται κάτι όμως που δεν γίνεται εύκολα. Οι πολίτες δεν ε, ενθαρρύνονται να το κάνουν εκτός και αν υπήρχε κάποιο χρηματικό αντίτιμο. Αν και αυτό επίσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε κερδοσκοπικά φαινόμενα, φαινόμενα κερδοσκοπίας μάλλον. Δύσκολο να βρούμε τη σωστή απάντηση, πρέπει όμως να το συζητήσουμε. Γι' αυτό θα δώσω το λόγο στην επόμενη ομιλητριά μας, την κυρία Γεωργία Δημητροπούλου, που έχει συντάξει μελέτη για τα θέματα της ε, επιμέλειας επιτροπίας, ε, guardianship, και θα μας μιλήσει για τα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ τα επόμενα 15 λεπτά θα προσπαθήσω να σας δώσω μια επισκόπηση της, ε, ε, των συστημάτων επιτροπίας και επιμέλειας στα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της στρατηγικής για την καταπολέμηση της εμπορίας και προκειμένου να υπάρξει μια κοινή κατανόηση για την επιτροπία και την εναρμόνιση των συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα... Το σύστημα είναι πολύ ευρώ και καθορίζει τα εθνικά συστήματα, τον διορισμό των ε, κυδεμών στα διάφορα κράτη-μέλη και τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν. Επικεντρωθήκαμε στο πώς οι εθνικές διατάξεις για την Επιτροπή εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται, στην περίπτωση αλλοδαπών ε, ανηλικών, θυμάτων εμπορία που δεν είναι απαραίτητος ε, υπήκοοι κάποιας χώρας, αλλά ε, παιδιά που βρέθηκαν μόνα τους σε μια άλλη χώρα σε κατάσταση κινδύνου και θα μπορούσαν να είναι θύματα εμπορίας. Πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου ότι τα παιδιά μπορεί να έχουν πέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης από εγκληματίες. Πολλοί από αυτούς ε, είναι πολλές φορές Ευρωπαίοι πολίτες. Προσπαθούμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται και σε αυτές τις περιπτώσεις. να ξεκινήσω στεκόμενοι σε ένα θέμα ορολογίας. Δεν υπάρχει γενικός αποδεκτός όρος για τον guardians ή guardian στον ευρωπαϊκό νόμο. Ο όρος χρησιμοποιείται και μεταφράζεται διαφορετικά με τρόπο ασυνεπή, ε, ε όχι συστηματικό. Οπότε Μπορεί να είναι ένα άτομο που περιγράφει νομοθεσία ως υπευθύνους, δαιμόνες προστάτες. Είναι τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι φροντίζουν ένα παιδί και είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Γενικώ μιλώντας υπάρχουν δύο κατηγορίες, δύο μάλλον ε, λογιών ε, ε, ε, ε, ευθύνε είναι ο νομικός εκπρόσωπος και ο κηδεμόνας. Οι νομικοί εκπρόσωποι, σε αντίθεση με τους επιτροπούς κηδεμόνες, έχουν πολύ περιορισμένα καθήκοντα που ορίζονται πολύ επακριβώς από τον νόμο ή βάση ή αναπερίπτωση. Και έχουν την ευθύνη να συνοδεύουν τα παιδιά σε συγκεκριμένε νομικέ διαδικασίε όπω τι αιτήσει ασύλου ή σε περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ε, παιδιών ε, ή σε περίπτωση που υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, εκεί πρέπει οι εκπρόσωποι να συνοδεύουν τα παιδιά στις νομικές διαδικασίες. Η διάρκεια της ευθύνης αυτής, του λειτουργήματος αυτού, λίγη οπότε ορίζεται. Ο κηδεμόνας ε, ξεπερνά τα στενά όρια της νομικής εκπροσώπησης, είναι κάποιο που ασχολείται με την υγεία και το καλύτερο συμφέρον, το μέγιστο συμφέρον του παιδιού σε όλε τι φάσει τη ζωή του, τη στέγαση, την υγεία, την κοινωνική του ζωή. Στην πράξη, σε εθνικό επίπεδο, βλέπουμε ότι τα δύο αυτά λειτουργήματα και καθήκοντα μπορεί να είναι διακριτά. Το βλέπετε ποιο είναι ο ρόλο του και στην πράξη Η νομική εκπροσώπηση είναι κάτι διαφορετικό. Κάποιες φορές υπάρχουν ε, δύο διαφορετικοί άνθρωποι που ασχολούνται με το ίδιο πεδίο, ένας ως νομικός εκπρόσωπο, ο άλλος ως κυδεμόνα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου χρειάζονται δικές γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη λόγω χάρη στι περιπτώσει των ετούντων άσυλο ή των θυμάτων εμπορία. όπου υπάρχουν περίπλοκες ποινικέ διαδικασίε. Οπότε ο κυδεμόνα δεν μπορεί να εξασκήσει καθήκοντα νομικό προσώπου, γι' αυτό διορίζεται ξεχωριστά νομικό εκπρόσωπο. Σε εθνικό επίπεδο σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν διατάξεις στην Εθνική Νομοθεσία για το διορισμό ενός κηδεμόνα. Εδώ λοιπόν οι κυδεμόνε αναλαμβάνουν γονικά καθήκοντα κάποιε φορέ σε περίπτωση που υπάρχει κάποια βία, περίπτωση βία, ε, ενδοκογενειακή βία, το παιδί πρέπει να βρεθεί υπό τη φροντίδα κάποιου, ασχολούνται και με τέτοιε περιπτώσεις. Οι διατάξει αυτές αφορούν όλα τα παιδιά και δεν αποκλείουν τα αλλοδαπά παιδιά, τα παιδιά που δεν είναι πολίτε μια χώρα. Η διαφορά είναι όμως ότι το καθεστώς ως προς τη διαμονή ενός παιδιού στη χώρα καθορίζει και την κυδαιμονία ή την επιμέλεια και είναι κρίσιμη σημασία στη δίκη υπηκότητα του παιδιού, αν είναι ε, παιδί της Ευρώπης ή από αλλού. Στις περισσότερες περιπτώσεις πέραν του νόμου για την προστασία των παιδιών και την ε, επιμέλεια και δαιμονία, υπάρχουν διατάξει στο μεταναστευτικό δίκαιο, το δίκαιο περί που, αφορούν και, που αφορούν και την νομική εκπροσώπηση. Οπότε στην πράξη τα ασυνόδευτα έχουν και νομικό εκπρόσωπο ή βάσει των διατάξεων του αστικού οικογενειακού δικαίου έχουν και κυδεμόνα εφόσον τους δοθεί διεθνής ε, προστασία. Αυτό και στα θύματα εμπορίας, εφόσον έχουν τακτοποιηθεί ασχέτως υπηκότητα. Τα περισσότερα κάτι μέλη τα εντάσσουν στη δική τους νομοθεσία περί προστασίας των παιδιών. τα παιδιά της Ευρώπης, τα παιδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρή πρόκληση και ε, ασυνέπειες ως προς την μεταχείριση που επιφυλάσσεται σε αυτά τα παιδιά στα διαφορα κατημέλη. Εάν εφαρμόζονται οι κανόνες ε, των ευρωπαϊκών κρατών ή όχι, γιατί σε καποια κατημέλη δεν ε, ισχύουν οι κανονισμοί μας ως νομικό εργαλείο, ιδίως σε περιπτώσεις απαγωγής ή καζόμενης εμπορίας, ή εφόσον κάποιο παιδί έχει υποχρεωθεί σε εγκληματικέ ενέργειε. Σε αυτέ τι περιπτώσει αποστέλλεται στο κράτο μέλο ε, τη ε, υπηκότητά του βάσει τη αστυνομική και δικαστική συνεργασία και των δικτύων τη ή μέσω πρεσβεία και δεν αναλαμβάνεται καμία δράση για το παιδί αυτό. Οι διαδικασίε διορισμού. Στα περισσότερα κράτη-μέλη, οι δικαστικές αρχές, αλλά σε άλλες περιπτώσεις διοικητικές αρχές, εφόσον αυτοί ορίζουν τον επιμελητή, διορίζουν όσο το δυνατόν συντομότερα, σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο σε κάποιες φορές ε, βάσει της νομοθεσίας. Όταν το χρονικό πλαίσιο προβλέπεται, ε, φτάνει και τις 8 μέρες, αλλά αυτό είναι έκτακτη περίπτωση. Σε πολύ λίγα κάτι μέλη βρίσκουμε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Οι διαδικασίες διορισμού ε, προβλέπουν ε, να αποφασίζει δικαστήριο, αλλά μπορεί να είναι και διοικητική αρχή. Λόγω χάρη στις κάτω χώρες, η αρχή για την ε, κυδαιμονία αναλαμβάνει την της κυδαιμονία του παιδιού στην περίπτωση τον Αγγλίκων αυτομάτως, με το που θα πατήσει ένα παιδί το πόδι του στη χώρα. Αυτό κάνει τα πράγματα να είναι λίγο πιο, τις λίγο πιο γρήγορες. Αλλά σε όλα τα κράτη-μέλη οι κατεπήγουσες περιπτώσεις καλύπτονται από προσωρινές επιτόπιες διευθυντήσεις για την επιμέλεια. Αυτές απαντώνται σε όλα τα κατημέλη και λόγω χάρη προβλέπουν και δαιμονία επιμέλειας τον χώρο υποδοχής του παιδιού, εκεί που θα βρεθεί και θα καταφύγει φτάνοντας σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Ελλάδα. Η ε, προσωρινά έχει ανατεθεί στον τοπικό εισαγγελέα. Στην πράξη, οι διατάξεις αυτές ισχύουν για να καλύπτουν τις επίγουσες ανάγκες νομικής εκπροσώπησης παιδιού, αλλά μπορεί να λάβουν μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό έχει ένα αντίκτυπο και στην ποιότητα των υπηρεσιών, διότι αυτοί οι προσωρινοί είναι ηλικιωμένοι σε πολλέ περιπτώσει και δεν έχουν και την εμπειρογνωμοσύνη για να φέρουν ει τα καθήκοντα τη κυδαιμονία τη επιμέλεια. Σε κάποιε χώρε υπάρχει ένα ειδικότερο σύστημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανάγκη αυτή να λάβουμε υπόψη μα τα ασυνόδευτα ανήλικα, όπως στις κάτω χώρε όπου υπάρχει ειδική αρχή, ή στο Βέλγιο, αλλά και στη Δανία. Υπάρχουν ειδικέ διατάξει για του ασυνόδευτου ανηλίκου. Η Εθνική Νομοθεσία για την Κυδαιμονία Επιμέλεια πολλές φορές προβλέπει οι συγγενείς, Η μέλη της οικογένειας να γίνονται κυδαιμόνες. Όταν όμως μιλάμε για συνόδευτα ενήλικα, μάλλον είναι απίθανο να υπάρχουν μέλη της οικογένειας ε, κάπου κοντά. Όταν τα παιδιά συνοδεύονται από ενηλίκους είναι διαφορετικά τα πράγματα. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Η μεγάλη δυσκολία είναι να καθοριστεί πρώτα απ' όλα η οικογενειακή σχέση με τους ε, ενηλίκους, αλλά εξίσου δύσκολο είναι να καταλάβει κανείς την ποιότητα της σχέσης με το παιδί. Μπορεί να είναι μια σχέση εκμετάλλευσης ή να υπάρχουν ε, δυσκολίες ε, στα σύνορα μέχρι να καταγραφεί η ταυτότητα του παιδιού. Δεν υπάρχουν λοιπόν πάντα τα εργαλεία εμπειρογνωμοσύνη για να αποτιμήσει κανείς τις σχέσεις, τους οικογενειακούς δεσμούς και πολλές φορές υπάρχουν τα λεγόμενα χωρισμένα παιδιά. Τα εγκαταλελειμμένα, αυτά που εγκαταλείφθηκαν τη στιγμή που πάτησαν το πόδι τους ένα κάτω από τον, ανήλικο, από τον ενήλικο που τα συνόδευε. Οι συνοδοί κάποιες φορές μπορεί να διοριστούν ως νομικοί πρόσωποι ή κηδημόνες του παιδιού εφόσον αποτιμηθεί η σχέση, αλλά παρόλα αυτά γίνεται πολύ δύσκολο να εντοπιστεί αν μιλάμε για περιπτώσεις αποπλάνησης, εκμετάλλευσης ε, ή οποιοδήποτε άλλη οποιοδήποτε άλλη μορφής βίας κατά του παιδιού. Κάτι άλλο σημαντικό, Πρόεδρε, κάτι που σήμερα παλεύουν να το λύσουν τα κρατημέλη, είναι το καθεστώς των κυδεμόνων. Θα πρέπει να είναι θελοντές, επαγγελματίες και τι είναι το καλύτερο για τα παιδιά. Η κυδαιμονία και η επιμέλεια έχει διοργανωθεί διαφορετικά στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κράτη όπου οι κυδαιμόνε είναι απλώ εθελοντέ, αλλά υπάρχουν και χώρε όπου οι κυδαιμόνε μπορεί να είναι και εθελοντέ και επαγγελματίε ή freelance. Όλε οι δυνατότητε υπάρχουν. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία όπω προκύπτει την έρευνά μα. Τι είδου κυδαιμόνα θα είναι τι σχέση θα έχει δηλαδή με τι αρχέ. Αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι τα προσόντα που διαθέτει ο κυδεμόνας. Και αν παρακολουθείτε η σχέση του με το παιδί και τι υπηρεσίε στήριξη υπάρχουν για να μπορέσει να φέρει πέρα στα καθήκοντά του. Τα καθήκοντα του κυδεμόνα επιμελητού είναι επίσης δύσκολα, διότι από τον νόμο δεν καθορίζονται σαφώς είναι ευρύτατη η εντολή που ανατίθεται σε ένα να Μπορεί να ασχοληθεί με την ευμερία του παιδιού ή γενικότερα να υποστηρίζει το παιδί, αλλά σε λίγε περιπτώσει υπάρχουν συγκεκριμένοι ορισμοί στην εθνική νομοθεσία. Μερικέ φορέ άλλα έγγραφα δίνουν κάποιες συστάσεις για το πώς θα πρέπει να φέρουν ει πέρα στα καθήκοντά του οι κεδεμόνες, αλλά δεν είναι νομικώ δεσμευτικά. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα είναι ότι στην πράξη η κυδαιμονία επιμέλεια είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται πολύ διαφορετικά μεταξύ των κρατών μελών και μάλιστα και εντός των κρατών μελών υπάρχουν σοβαρές διαφορές. Πολλές φορές υπάρχουν και θετήσεις σε τοπικό επίπεδο, οπότε οι πρακτικές των είναι τελείως διαφορετικές. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα για την διαδικασία αποτίμησης της ηλικία. Αυτό έχει γίνει προσπάθεια να καλυφθεί και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά πολλές φορές οι κηδεμόνες ορίζονται μετά το τεστ. Και όχι πριν. Εδώ ε, για τα ε, ασυνόδευτα, όπως έλεγα προηγουμένως, το ανέφεραν και οι προηγούμενοι, το δίκαιο για τη μετανάστευση και το άσυλο υποτίθεται ότι προστατεύει το μεγαλύτερο συμφέρον, το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. Αλλά εδώ υπάρχουν συνέπειε ε, στην πράξη και εφόσον υπάρχει κατακαιρματισμό και ασυνέπεια στην πράξη, το δίκαιο δεν λειτουργεί. Δηλαδή, Πραγματικά το καθεστώς του παιδιού προς τη διαμονή καθορίζει τελικά και τη φροντίδα και την, ε, το είδος και δαιμονίες επιμελίας που θα λάβει. Μια άλλη από τις βασικές δυσκολίες είναι οι καθυστερήσει στο διορισμό των επιμελητών επιτρόπων. Αυτέ ε, οφείλονται σε διαφορετικού λόγου, λόγω χάρη στι ε, δικαστικέ διαδικασίε που μπορεί να διαρκούν πολύ, να διονύζονται. Μια άλλη σημαντική κουβέντα είναι η διαδικασία καταχώρησης των ε, παιδιών που ξεκινάει στις υπεύθυνε υπηρεσίες και αναφέρθηκε ήδη το θέμα της αποτίμησης της ηλικία. Δεν υπάρχει αναρμονισμένη διαδικασία εδώ. Στην πράξη Η ε, διαδικασία αποτίμησης της ηλικία για θέματα ασύλου μπορεί να διαφέρει από την ποινική διαδικασία στο ίδιο κράτος μέλος ή μεταξύ ε, της διαδικασίας που υπάρχει για τους δράστες και για τα θύματα σε ποινικέ διαδικασίες. Σοβαρές ε, ή για το πώς τεκμηριώνεται η αποτίμηση της ηλικία είναι και αυτό ένα θέμα. Η τεκμηρίωση δεν είναι πάντοτε υποχρεωτική. Τα θέματα αυτά λαμβάνουν νέα σημασία όταν μιλάμε για συνόδευτους ανηλίκους, διότι στις διαδικασίες καταγραφής του παιδιού, στις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως στις περιπτώσεις ασύλου, είναι ένα θέμα πώς καταγράφονται τα δεδομένα στο Eurodac. Εάν τα δεδομένα μπουν στο Eurodac ή στη βάση δεδομένων της αστυνομίας, μετά δεν αλλάζουν και αυτό έχει σοβαρότατα αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών έχει νομικές συνέπειες. Γιατί τα δεδομένα που έχουν σε αυτές τις νομικές βάσεις δεν αλλάζουν. Επίσης μια άλλη δυσκολία είναι να εντοπιστεί το καθεστώς του παιδιού, η κατάσταση του παιδιού ως προς το ασυνόδευτο ή όχι. Για πολλά παιδιά τα συνόδευτα έχουμε διαφορετικές ε, διαδικασίες. Ε, για παράδειγμα, μπορεί να βρεθούν ανήλικα παντρεμένα και ο ενήλικος που είναι ο σύζυγος ή σύντροφος να οριστεί και μόνος συνομικός εκπρόσωπος. Εκεί δυσκολεύονται πάρα πολύ τα, πράγματα, πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί οι αρχές για την προστασία των παιδιών πώς θα αποτιμήσουν τη σχέση αυτή. Είναι, είναι καταναγκαστικός ο γάμος, είναι περίπτωση εκμετάλλευση του παιδιού. Δεν είναι δυνατόν να ισχύσουν όλα αυτά και χάνεται το συγκεκριμένο παιδί. Και κάποια στιγμή διορίζεται ένας προσωρινός κυδεμόνας ώστε μακροπρόθεσμα να μπορέσει να αποτιμήσει τη σχέση με το παιδί και να δει την ποιότητα της σχέσης αυτής του δεσμού ε, εξατομικευμένα. Τέλος, ήθελα να θέσω το θέμα της διεθνούς συνεργασίας. Σε όλε τι περιπτώσει προστασία των παιδιών, αλλά ιδίω ό,τι αφορά την εμπορία των παιδιών, την επανένωση οικογενειών και όσα εμπίπτουν στον γενικανισμό του Δουβλίνου. Ο ρόλο των κυδεμόνων εδώ είναι πολύ περιορισμένο. Διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ νομίζω Οι δαιμονές δεν έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Κάποιες φορές συμμετέχουν στις διαδικασίες, διότι πρέπει να διασφαλίσουν το καλύτερο συμφέρον του παιδιού. Αλλά σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει πολύ συγκεκριμένο ορισμός για του δαιμόνες που θα πρέπει να κάνουν στις διάφορες διαδικασίες η αποτίμηση της σχέσης και του οικογενειακού δεσμού του παιδιού με τον ε, ενήλικο που το συνοδεύει ή με άλλα μέλη της οικογένειας που είναι μαζί ή έχουν μείνει πίσω στη χώρα τους είναι θέματα που, που διακανονίζονται στον κανονισμό του Δουβλίνου και αυτό είναι δύσκολο να το καθορίσουν και οι δαιμόνε, οι αρχέ που είναι υπεύθυνε για την ανάστευση. Οι αρχέ για την εξέταση τη αίτηση ασύλου λόγω χάρη μπορεί να ασχοληθούν με το θέμα αυτό ή οι αρχέ προστασία του παιδιού που έχουν την αρμοδιότητα και την εμπειρογνωμοσύνη να ε, αποφασίζουν για τέτοιε περιπτώσει. Νομίζω ότι το δίκτυο των Ευρωπαίων Guardian, ε, επιμιλητών και επιτρόπων, κυδεμόνων και επιτρόπων μάλλον, βασίζεται σε ένα επικαιροποιημένο κείμενο τη Επιτροπή που θέλει να δημιουργήσει ένα τέτοιο δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα συνέβαλε τα μάλα στην ενίσχυση τη διεθνού συνεργασία και τα θέματα αυτά να συζητηθούν με ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα τη κυδαιμονία. Δεν είναι σαφέ πότε λίγη η κυδαιμονία. Οι νομικέ διαδικασίε των κρατών μελών, όταν με δικαστική απόφαση διορίζουν τα κυδαιμόνα, δεν προβλέπουν ποτέ λίγη. Χρειάζεται δικαστική απόφαση για να λήξει η Και αυτό δημιουργεί δυσκολίε. Όταν τα παιδιά πρέπει να μεταφερθούν ε, έστω και από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Σα ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you, thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που άργησα. Παρ' όλα αυτά εντυπωσιάστηκα από τις παρουσιάσεις σας. Και τώρα ερχόμαστε στο γύρο των αρταπαντήσεων. Ευχαριστώ πολύ που μας ε, αναφέρατε όλες τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά την παιδική μέρημνα. Έχω ένα ευρύ ερώτημα διότι δυσκολεύομαι να καταλάβω, παραδείγματος χάρη, η σύμβαση για τα παιδιά, πώς εφαρμόζεται. Είμαι Δανός, μιλήστε για τη χώρα μου, γνωρίζετε ότι στη Δανία τα δικά μας παιδιά τα φροντίζουμε ιδιαιτέρως, αρκεί δηλαδή να έχουν τη δανική ποιότητα, όμως η κυβέρνησή μας δεν διστάζει να χωρίσει τις οικογένειες των μεταναστών, τα μέλη τους δηλαδή. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή στέλνουμε παιδιά πίσω στη Σομαλία, για να σας ένα παράδειγμα. Παιδιά όμως που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Δανία. είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω. Πότα, πρώτα, αυτή η σύμβαση για τα παιδιά πώς ισχύει έχει, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Τι πρέπει να προσθέσουμε ώστε να υπάρχει η εξασφάλιση της ε, ελάχιστης ε, δίκης μεταχείρισης του παιδιού και ισότητας μεταχείρισης. για μη παιδιά που δεν, έχουν, που δεν είναι παιδιά Ευρωπαίων μιλάω. Αν κερδίσει η Μέρκελ στις γερμανικές εκλογές, μπορεί να μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στη συνθήκη. Εμείς ως πολιτικοί τι πρέπει να κάνουμε, ώστε όλα τα παιδιά που ζουν στην Ευρώπη ε, να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Πώς θα ισχυροποιήσουμε τα δικαιώματά τους. Και σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της δικαστικής, δεν ξέρω αν μου απαντήσετε βέβαια αλλά θα ήθελα έστω τη συμβουλή σας. Είναι δύσκολο το ερώτημα και δεν νομίζω ότι είμαι και εγώ η καταλληλότερη για να απαντήσω. Αλλά ακούγοντάς σας ε, σκέφτηκα το εξής. Το βασικό πρώτα απ' όλα είναι η εθνική νομοθεσία σε ό,τι αφορά το εθνικό δίκαιο περί και περί μετανάστευσης ε, να ε, είναι εναρμονισμένο. Και αυτή είναι αφετηρία. Δεν είναι ναι, ισχύει μόνο για τη Δανία. Πρέπει να δούμε ο καθένα τη χώρα μα και να δούμε την νομοθεσία για την παιδική μέρη και τη μετανάστευση και να δούμε τι ασυνέπειες υπάρχουν και να άρουμε αυτές τις ασυνέπειες. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί η εθνική νομοθεσία περί παιδική μέρη για αυτά τα παιδιά, για την Επιτροπή για παράδειγμα που προτεραιότητα σε όλες τις χώρες δίνεται στο διορισμό των μελών της οικογένειας, των συγγενών, που είναι και λογικό, γιατί έχει κάποιον οικογενειακό δεσμό ήδη, το άτομο με το παιδί. Και είναι το καταλληλότερο για να έχει το ρόλο του μόνο. Αλλά θα πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχουν πάντα οι καλές γιαγιάδες ε, που θα αναλάβουν το παιδί αν έχουμε ένα παιδί που δεν ξέρω από πού μπορεί να έρχεται, Σομαλία, Ιράκ, Συρία κτλ. κτλ και το συνοδεύει κάποιο που δεν ξέρει ποιο είναι τελικά, εκεί όταν εφαρμόζουμε αυτές τις διατάξεις θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να τι εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αξιολογήσουμε τη σχέση ένα παιδί που ε, δεν μπορεί να αποδείξει τη σχέση την οικογενειακή, ε, πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, την ε, ασυνέπεια που υπάρχει κατά πολέμηση διακρίσεων, αυτά. Πρόεδρος, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να απαντήσει στο ερώτημα αυτό, όμως έχω και ένα κύριο εκεί πίσω που ζήτησε το λόγο. Αλλά πρώτο κύριο Σφανλό, Για να προσπαθήσω να απαντήσω. Εσείς φαίνεται να λέτε ότι δεν υπάρχουν ε, ένδικα μέσα. Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Πώς θα εφαρμόζουμε το θέμα. Έχουμε τη, παιδική, τη σύμβαση για τα παιδική μέρηνα και στο άρθρο 3 λέει ότι πρέπει να κατησχύει το συμφέρον του παιδιού. Είναι δύσκολο, κάτε με, να πει κανεί ότι ένα παιδί που γεννήθηκε στη Δανία, έχει ζήσει στη Δανία, οι φίλοι του μιλάνε Δανέσκ κτλ. κτλ ότι αυτό το παιδί μπορείτε να το στείλετε που το είπατε, που είπατε στη Σομαλία, στην Ιγύρια, τέλο πάντων. Και να πει κανεί δε ότι είναι και προ το συμφέρον του κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί και στη Δανία ένα τρόπο. ίσως με δικαστικές διαδικασίες και ίσως με τη βοήθεια των ΜΚΟ, ώστε να εφαρμοστούν οι ισχύοντες νόμοι. Δεν είναι και τόσο τραγικό. Ε, μπορεί να γίνει, χρειάζεται δράση. Σε κάποιες χώρες ε, στην Ευρώπη είναι προφανές ότι δεν προτατήλησε ένα παιδί υπό αυτές τις συνθήκες πίσω στη Σομαλία, για παράδειγμα. Τα λέει και η σύμβαση για τα δικαιώματα των παιδιών. Το θέμα είναι πώς θα εφαρμόσουμε καλύτερα τους ενισχύ νόμου. Και όχι να προσθέσουμε νέα στρώματα. Already, Δεν ξέρω να συμφωνούν και οι συνάδελφοί μου. Να δώσω στον κύριο. Δώσω λόγο στον κύριο εκεί στο βάθος παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Φίλιππε Λορτή, πρώτος γραμματέας της διάσκεψης της Χάγης ε, για το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο. Η διάσκεψη της Χάγης ε, καλωσορίζει τις μελέτες αυτές ε, που παρουσιάστηκαν και συμφωνούμε με κάποια από τα ευρήματα. Ε, Βεβαίω έχουμε και την μελέτη για την εφαρμογή της σύμβασης του 1996 αυτή η μελέτη διεξάγεται σε συνεργασία με τη UNICEF, την υπατερμοστία του ΕΕ, για τους πρόσφυγες, την Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία και την ε, Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η τελευταία αυτή η επιτροπή στο Γενικό Σχόλιο Υπαριθμών 5 του 2005 πρότεινε την ε, εφαρμογή της Σύμβασης του 96 σε αυτόν τον τομέα και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατευθυντήρες γραμμές ε, για την εναλλακτική κυδαιμονία ζήτησε από τα κράτη να εφαρμόσουν τη Σύμβαση του 1996 για τα συνόδευτα ανήλικα. Συμφωνούμε με τη μελέτη, με την έννοια ότι ο όρος ταραχές πρέπει να ερμηνευθεί ευρεία τη ενία. Αυτό συμφωνεί με το Γενικό Σχόλιο Υπαριθμών 5 του ΟΗΕ, παραγράφους 84-88, περιλαμβάνει πίνες, ε, λιμούς, με συγχωρείτε, εμφυλίους πολέμους, καταστροφές και κοινωνικο-οικονομικές τάραχες. Συμφωνούμε με την έννοια ότι ο κανονισμός των Βρυξελών 2α στην Ευρώπη, όπως φαίνεται, θα καλύπτει μόνο παιδιά από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία γιατί το άρθρο 61 προβλέπει ότι ο κανονισμός ισχύει μόνο για παιδιά τα οποία είναι κάτοικοι της Ένωσης. Επίσης, συμφωνούμε ότι η αρχή της σύμβασης του 1996 είναι πιο εξελιγμένη από τον κανονισμό Βρυξέλλες Ιόλφα. Επίσης, συμφωνούμε πλήρω πώ η Σύμβαση του 1996 δεν περιορίζεται στην εφαρμογή της με τα άλλα συμβαλώμενα μέρη. Υπάρχουν ε, οι κανόνες ε, περί δικαιοδοσίας, το άρθρο 13 του Βρυξελών 2α είναι το άρθρο 6 του δικού μας και ισχύει ανεξαρτήτως του εάν το παιδί έχει τόπο συνήθως κατοικία σε συμβαλώμενο μέρος ή όχι. Το ίδιο ισχύει και για τα άρθρα 11 και 12. Και αυτά ισχύουν για το τι γίνεται όταν ένα παιδί επιστρέφεται σε μη συμβαλόμενο κράτος. Όμως, με τα μη συμβαλόμενα κράτη δεν ισχύει αυτό το σύστημα, αλλά αυτό το οποίο γνωρίζουμε από την πράξη της Τσεχίας, παραδείγματος χάρη, είναι ότι τα κράτη συνεργάζονται με τις ε, ε πρεσβείες αυτών των χωρών και τα προξενία αλλά και με τον Ερυθρό Σταυρό και την οργάνωση Save the Children για να σταλούν τα παιδιά αυτά σε μη συμβαλόμενες χώρες. Έχουμε νομολογία από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 11 σε μη συμβαλόμενα κράτη. Αυτό πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει. Τα παιδιά λοιπόν αυτά είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και απαιτείται μια παγκόσμια λύση και αν θέλουμε να έχουμε ίση μεταχείριση για όλους τους ανηλίκους ε, κατά την άποψή μας θα πρέπει να ε, ισχύσει η σύμβαση του 1996. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που διαβάζουμε στη μελέτη ότι υπάρχει μια σύσταση που λέει ότι όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να προωθήσουν παγκοσμίω τη σύμβαση του 1996. Να πάμε ακόμα παραπέρα και να ζητήσουμε την παγκόσμια εφαρμογή της σύμβασης του 96 σε αυτόν τον τομέα. Να απλουστεύσουμε την ζωή των διακινητών και να τους πούμε ότι υπάρχει μόνο η σύμβαση του 96. Αντί ε, να έχουμε δηλαδή ενιαίους κανόνες και θα θέλαμε να υπάρχει να υπάρχουν ενιαίου κανόνες και, ενιαίοι κανόνες και για τους ασυνόδευτούς ανηλίκους. Και εδώ πέρα μας στηρίζει και η UNICEF και η Πατερμοσία του για τις πρόσφυγες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και για την παρέμβαση αυτή, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι θέλουν να αντιδράσουν ε, σε, αυτή την, ε, σε αυτό το σχόλιο. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, αλλά επανέρχομαι σε εσά κύριε μου. Διότι εγώ δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι πρέπει να δούμε την νομική βάση σε ό,τι αφορά την παιδική μέρημνα, διότι... Διότι λέγω, στη Δανία για παράδειγμα, δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο όταν η κυβέρνηση, οι αρχές αποσπούν ε, το παιδί από την οικογένειά του. Μόνο διοικητικές ε, μπορεί να είναι οι προσφυγές. Και όποτε έρχομαι σε επαφή με το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και του αρμόδιου για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτρόπου μου λένε ότι δεν είναι καθόλου σαφές αν αυτό είναι εντάξει ή όχι. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επιληφθεί τέτοιων υποθέσεων. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω πολλούς από τους ανθρώπους αυτούς, από αυτές τις οικογένειες και πολλές φορές μου λένε πρόσεχε πάρα πολύ. Γιατί μπορεί το δικαστήριο να μην επιληφθεί καν. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είναι σαφή η νομική βάση. Γιατί αν οι ειδικοί δεν μπορούν να μου ξεκαθαρίσουν εμένα αν αυτή η υπόθεση είναι καλή ή κακή, νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη νομική βάση. Αν μου επιτρέπετε να απαντήσω, μιλήστε για το δικαστήριο του Στρασβούργου και το ρόλο του. Αυτό είναι άλλο. Είναι δύσκολο θέμα. Δεν είναι αρμόδιο το δικαστήριο για θέματα ασύλου. Έχουν πάρει τι αποστάσει του από αυτά τα θέματα. Είπατε όμω ότι στη Δανία είναι δύσκολο τα δικαστήρια να ασχοληθούν. Μήπω αυτό λοιπόν είναι πρωταρχικό καθήκον των αρχών στη Δανία. Είναι τέτοια στερική δομή που έχει αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή να είναι δυνατόν να λειτουργήσουν τελικά οι ευρωπαϊκοί διεθνείς κανόνες. The... Νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά έχετε εντοπίσει είναι μια έλλειψη του δανέζικου συστήματος και δεν είναι ελάττωμα του διεθνούς δικαίου. Αλλά και πάλι θα θέλω να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων μου. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τους εμπειρογνώμονές μας ίσως. Αν θέλει κάποιος να αντιδράσει, αλλά όχι μόνο για τη Δανία. Να πολύ να πω λίγο κάτι. Για μένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ανηλίκων είναι παγκόσμια. Δεν είναι θέμα λοιπόν δανέζικου δικαίου. Εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε στο διεθνές πλαίσιο και μια διεθνή νομική βάση κατά την άποψή μου και εκεί λέτε ότι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν είναι αρμόδιο να δει τις περιπτώσεις ομαλών ενώ είναι Το έχουμε κάνει, έχουμε πάει στο δικαστήριο το 2013, το 2015 και το 2011. Οπότε υπάρχει κάποιο δεδικασμένο. Γι' αυτό ε, ερωτώ, ε, γιατί δεν είναι σαφές ε, και οι απαντήσεις που λαμβάνω είναι επίσης ασαφείς. Λοιπόν, αν να έχουμε μια παγκόσμια φροντίδα παιδιών, Μήπω η απάντηση είναι ε, μια καλύτερη διεθνή νομική βάση. Μάλιστα. Όχι, ε, μπορεί να χρειάζεται βελτίωση νομοθεσία, αλλά σε γενικές γραμμές ε, νομοθεσία υπάρχει. Υπάρχει θέμα ασυνέπειας μεταξύ διαφορετικών νομοθετημάτων κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να διαλέξουμε τι θα εφαρμόσουμε, π.χ. για επιστροφές και επιστρέφεται και ε, καλώς επιτρέπεται γιατί σε κάποιες περιπτώσεις καλό είναι ένα παιδί και λογικό να, να μην ξαναπάει στη χώρα προέλευσης γιατί έχουμε περιπτώσεις ε, οικογενειακής ε, πανένωσης ή είναι προς το συμφέρον του παιδιού αλλά Υπάρχουν και άλλες απαιτήσει μετά για να υπάρχει κάποια επιστροφή. Οπότε, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς εφαρμόζονται αυτά και ποιος κρίνει. Θα επιμείνω εγώ σε αυτό. Νομίζω πως όλες οι παρουσιάσεις ε, αναφέρουν πως ε, υπάρχει περιορισμένος ε, ρόλος ε, των ε, αρχών προστασίας των ε, παιδιών. Οπότε το αναλαμβάνονται οι αποφάσεις αυτές από του αρμοδίους μετανάστες. Δεν είναι θέμα αν είναι καλοί ή κακοί άνθρωποι. Μπορεί να μην έχουν την σωστή κατάρτιση αν ήμασταν στη Δανία, στην Ελλάδα, κανείς δεν σκεφτόταν ε, ο αστυνομικό ή κάποιο από τον τομέα της μετανάστευσης να κρίνει το συμφέρον του παιδιού. Θα είναι οι, οι αρχές που κρίνουν για τους ανηλίκου. Τον μιλάμε δηλαδή για τους κηδεμόνες ε, γενικά προβλέπεται ότι θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Όταν μιλάμε λοιπόν για τις διαδικασίες επιστροφών, είναι ε, δυνατόν να υπάρχει αξιολόγηση πως ε, δεν θα πρέπει να μπλοκαριστεί η διαδικασία. Όχι. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια αρμοδιότητα. Στην Ολλανδία υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις όπου τα εθνικά δικαστήρια αναγνώρισαν πως οι αρχές δαιμονία είχαν την ε, εμπειρογνωμοσύνη να αποφασίσουν το συμφέρον του παιδιού. Αλλά αυτό είναι μια νέα εξέλιξη. Αλλά δεν έχουν αρμοδιότητες, ποιο το νόημα. Οπότε πρέπει να δούμε αν έχουν και την δυνατότητα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ε, κατά την άποψή μου δεν είναι έτοιμη. Και στις περιπτώσεις ε, που αντιμετωπίζουμε αυτό δεν γίνεται πάντα αποτελεσματικά γιατί υπάρχουν ζητήματα γλώσσας, ε, πολιτισμού, διάφορα γραφειοκρατικά και επί, χωρίς απαραίτητους πόρους δεν θα μπορέσουν και σε πολλές χώρες, δεν θέλω να πω σε όλες, γιατί αναφέρθηκε και η Τσεχία που υπάρχει η κεντρική αρχή με 50-70 άτομα προσωπικό που είναι πολύ ε, καλό παράδειγμα του πώς πρέπει να αναπτύσσονται οι κεντρικές αρχές. Μετά έχουμε χώρες όπου η κεντρική αρχή είναι ένα άτομο που κάθεται σε ένα υπουργείο, στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Ε, ε, κοιτάζει χαρτιά. Λοιπόν, ε, αυτά είναι ζητήματα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει είναι αυτή η πρόταση. Αλλιώς ε, δεν μπορούμε να μιλάμε για εφαρμογή στην πράξη. Αυτή είναι η άποψή μου. Maybe Απλώς να προσθέσω ένα παράδειγμα. Το θέμα δεν είναι να έχουμε νέους κανόνες, αλλά να εφαρμόσουμε αυτούς που υπάρχουν. Οι μεταφορές βάσει του Δουβλίνου. Όταν ένα παιδί ξέρει ότι κάποιο τέλο πάντων, ή ο δεν ή οι αρχέ, βρήκαν μέλη τη οικογένειά του, αλλά κάποιο μέλο γίνεται αίτηση για μεταφορά. Ξέρω εγώ η μητέρα να πάει από την Ελλάδα στη Γαλλία για το παιδί. Και εντό αυτού του πλαισίου υπάρχει ο κανονισμό του Δευλίνου. Προβλέπει. Προβλέπει στο άρθρο 3 τη σύμβαση για τα παιδιά. Και τι συμβαίνει σε αυτέ τι περιπτώσει. Οι αρχέ, οι αρχέ μετανάστευση λαμβάνουν την απόφαση για τη μεταφορά. Οι ελληνικέ και γαλλικέ αρχέ, στην παραδείγμα μου. Και τις αποφάσεις αυτές τις λαμβάνουν στη διακριτική του ευχαίρεια βέβαια. Δηλαδή αν οι γαλλικές και ελληνικές αρχές αρνηθούν ξέρω εγώ τη μεταφορά του παιδιού εάν θεωρήσουν ότι δεν είναι προς το μέγιστο συμφέρον του παιδιού να βρίσκεται με τη μάνα του στον κανονισμό του Δουβλίνου δεν λέγεται πουθενά. Δεν διευκρινίζεται Δεν υπάρχει εργαλείο ή απόφαση των αρχών αυτών να ε, προσβληθεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης ε, να αμφισβητηθεί. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Μόνο οι αρχές αποφασίζουν. Δεν υπάρχει δικαστική διαδικασία, οπότε τα εργαλεία υπάρχουν μεν. Τα ένδικα μέσα υπάρχουν, αλλά χρειαζόμαστε νομικές διαδικασίες. Να μπορεί να αποτιμηθεί και σε ένα σαφές νομικό πλαίσιο το μέγιστο συμφέρον του παιδιού. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει το άρθρο 3 και όλε οι αποφάσει θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέγιστο συμφέρον του παιδιού, αλλά αν δεν υπάρχει κανεί να το αποτιμήσει ή να αμφισβητήσει μια λάθο απόφαση, εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση και όχι να σκεφτούμε νέου κανόνε. Κάτι υπάρχει στον κανονισμό του Δουβλίνου θα μπορούσε να μα εξυπηρετήσει στα άλλα νομικά μέσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνεισφορά σας. Έχετε ζητήσει και εσείς το λόγο. Γεια σας, καλησπέρα. Ε, Κωνσταντσα Χέρμαν από το Ιταλικό Υπουργείο Δικαιοσύνη. Κάτι που ήδη θίξατε κάποιοι από εσά, αλλά ήθελα να επανέλθω. Ότι μάλλον δεν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω νομοθεσία, αλλά περισσότερο συντονισμό. Εγώ θέλω να τονίσω το εξή για του ασυνόδευτου ανηλίκου, τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Τι γίνεται με αυτά που δεν κάνουν αίτηση ασύλου τα κενά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία προφανώς είναι διαφορετικά. Πώς μπορεί το θέμα αυτό να καλυφθεί από το Διεθνές Ιδιωτικό Δίκαιο. Πρέπει εκεί να κάνουμε κάτι περαιτέρω. Γιατί στη δική μου τη χώρα οι ασυνόδευτοι ανήλικοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιστραφούν. Οπότε πρέπει να βρούμε ένα πάτημα, ένα νομικό πλαίσιο για αυτού όταν βρίσκονται στην Ευρώπη. Το ερώτημα λοιπόν είναι για αυτά τα παιδιά που δεν ζητούν άσυλο. Ναι, κέριο ερώτημα. Διότι είναι ένα μεγάλο αριθμό παιδιών αυτό, αυτά που δεν ζητούν ε, άσυλο που δεν εκπληρούν τι προποθέσει για να το επιθούν ή να πάρουν το καθεστώ του πρόσφυγα σε πολλέ χώρε. Στη Γαλλία, λόγου χάρη. Τα μία συνόδευτα παιδιά προστατεύονται κατά των αποφάσεων επιστροφή και απομάκρυνσης την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών, οπότε εκεί πρέπει να βρεθούν λύσει διαρκεία για τα παιδιά για να προστατευτούν. Ό,τι προβλέπεται αυτή τη στιγμή για τα παιδιά που αιτούνται άσυλο δεν ισχύει αυτομάτως και για αυτά που δεν το αιτούνται. Ένα παράδειγμα. Όλες οι δυνατότητες να ε, επανενωθεί το παιδί με άλλα μέλη της οικογένειάς του που βρίσκονται σε άλλα κάτι μέλη προβλέπεται το κανονισμό του Δουβλίνου απέναντίας δεν υπάρχει τίποτε εκτός Δουβλίνου για τα παιδιά που δεν ζητούν άσυλο. Υπάρχει η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης, αλλά αυτή προποθέτει ένα μέλος της οικογένειας, γονέας ή άλλο, διαμένει νομίμως σε άλλο κάτω μέλος. Πολύ συχνά αυτό δεν συμβαίνει. Μπορεί να βρίσκονται στην Ευρώπη άλλα μέλη της οικογένειας, αλλά δεν σημαίνει ότι το καθεστώς τους είναι νομικά ξεκαθαρισμένο, οπότε δεν ισχύει αυτό της οικογενειακής επανένωσης και δεν έχουμε και κανένα εργαλείο για τη μεταφορά του παιδιού, που να γίνει τουλάχιστον με τρόπο έφτακτο ακόμη και βάσει του κανονισμού Βρυξελών 2 ε, 2B δεν μπορεί να ε, τοποθετηθεί το παιδί σε άλλο κατός μέρος με τον πατέρα ή τη μητέρα, διότι δεν προβλέπεται αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πραγματικά κενά στην ισχύουσα νομοθεσία για αυτά τα παιδιά. Όντως. Ευχαριστώ. Η σύμβαση τη Χάγης θέλει το λόγο. Ναι, η διάσκεψη τη Χάγη. Όλε αυτέ οι βιώσιμε λύσει οι λύσεις διαρκεία, όντω, προβλέπονται στο πεδίο εφαρμογή τη Χάρτα το άρθρο 3. Οι μεταφορέ αυτέ οι τοποθετήσει, οι οικογενειακέ επανανώσει σε τρίτο κράτος, σε προέλευση ή σε τοπικό επίπεδο, καλύπτονται από τη σύμβαση του 1996. Οι κανόνε για τη διοικητική συνεργασία προβλέπονται εφόσον είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση της Χάκης του 1996. Μόνο οι λύσεις που δεν είναι δυνατή στη Σύμβαση του 1996 είναι η διεθνής υιοθεσία που καλύπτεται από άλλο εργαλείο το 1993. Όμως σας καλώ στο ιστότοπό μας ε, μέχρι το τέλος Ιουλίου να δείτε τη μελέτη που θα παρουσιαστεί. Γιατί όλες ε, οι περιπτώσεις καλύπτονται και θα έχουμε και ένα κατάλογο όλων των διατάξεων που είναι εφαρμοστές και πώς μπορούν, μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν αμφιβάλλω ότι η σύμβαση μπορεί να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα. Όμω, αν κατάλαβα καλά, το πρόβλημά μα είναι η εφαρμογή. Διότι ακόμα και μόνο ο όρο επί της αρχής ή καταρχήν είναι πολύ καλός όταν ακούγεται, αλλά το θέμα είναι πώς εφαρμόζονται τα πράγματα και στην πράξη. Θέλετε να αντιδράσετε κυρία μου, ναι. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι καλύπτονται όλα. Διότι να σα δώσω πάλι το παράδειγμα που έλεγα πριν. Ένα παιδί που δεν ζητά άσυλο και βρίσκεται στη Γαλλία και ο πατέρα του βρίσκεται στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διαδικασία τη τοποθέτηση που προβλέπει η Σύμβαση τη Χάγη, γιατί στο άρθρο 33 ε, γίνεται λόγο για τοποθέτηση του παιδιού σε οικογένεια υποδοχή σε ένα ίδρυμα, ούτε το ένα μας αφορά ούτε το άλλο, ανάλογο φορέα, ούτε αυτό ισχύει. Θέλουμε απλώ να πάει να βρει τον πατέρα του δεν προβλέπεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Υπάρχουν λοιπόν κενά. Και αυτή τη στιγμή η πρόταση του εισηγητού του Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της διαδικασίας των Βεξελών 2, bis, 2α, προβλέπει να αναθεωρηθεί η διαδικασία της τοποθέτησης σε αυτόν τον κανονισμό, ώστε να υπάρχει δυνατότητα το παιδί να πάει να βρει ένα μέλος της οικογένειάς του, κάτι που θα κάλυπτε καταστάσεις που τώρα δεν καλύπτονται. Είναι πολύ σημαντικό αν εγκριθεί αυτή η αναθεώρηση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο. Ναι, αλλά για να απαντήσω σύντομα, η μεταφορά αυτή δεν θα γινόταν βάση των κανόνων συνεργασία, αλλά βάσει των κανόνων δικαιοδοσία. Είναι δυνατόν να γίνει μεταφορά τη δικαιοδοσία βάσει των άρθρων 8 και 9 για να μεταφερθεί η δικαιοδοσία προ τη δικαιοδοσία που βρίσκεται ο πατέρα και ειλικρινώ, χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών για να εντοπίσουν του γονεί. Γονεί με του οποίου μπορεί να επανενωθεί το παιδί. Η διαδικασία μέσω μεταφορά τη δικαιοδοσία και όχι δικαστική συνεργασία. Να μια πληροφορία που πρέπει να την αφομοιώσουμε, να τη χωνέψουμε, να την ελέγχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ζητήσει κάποιο. Α, κύριο Ρόπ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις παρεμβάσεις σας. Σε ένα σχεδόν τέλειο κόσμο, η συζήτηση θα πρέπει να είναι τις συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα, πώς θα τα εφαρμόσουμε στην πράξη. Αυτή να βάλω και τα ακουστικά. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι παραβλέπετε παρόλα αυτά μια σημαντική λεπτομέρεια, ότι δηλαδή οι κυβερνήσει στην Ευρώπη θέλουν να προσβάλλουν την σύμβαση και όχι να την εφαρμόσουν. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε από κοινού. Εγώ το θεωρώ τεράστιο το πρόβλημα. Να έχουμε τις κυβερνήσεις πλούσιων χωρών να στοχεύουν συνεχώς, ή τόσο να λένε ότι θέλουν να προσβάλλουν τις συμβάσεις που έχουμε. Αυτό το πρόβλημα πώς θα αντιμετωπίζουμε. <laughs> oh, I'm sorry. Ε, συγγνώμη, ε, μα συγγνώμη, συγχωρείτε που μιλάω, κυρία Πρόεδρε. Όχι, όχι, καλά κάνετε, καλά κάνετε. Μας αρέσουν αυτά. Ε, γιατί κοιτάω εδώ πέρα τα πρόσωπα των ειδικών και δεν ξέρω σε ποιον, ε, να... σε ποιον απευθύνεται το ερώτημα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, αλλά έτσι όπως το διατυπώνετε, δείχνει ήδη ότι δεν είναι η νομοθεσία η απάντηση. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα, είναι το κράτος δικαίου και ε, άρα είναι εξόχως πολιτικό ζήτημα. Αυτό είναι μετά άλλο, άλλο παπά Ευαγγέλιο. Ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευρά νομική, αλλά κάποια στιγμή φτάνουμε στα όρια. Αν οι πολιτικοί δεν σέβονται τον νόμο, τι, τι να κάνει ο νόμος. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και πρέπει να υπάρξει πολιτική κινητοποίηση ακριβώ για να διατηρηθεί το κράτος δικαίου. Και αυτό συχνά κάνουμε. Ναι, ναι. Πρέπει ακριβώς να υψώσουμε το αναστημά μας για το κράτος δικαίου και να εφαρμόσουμε τις αρχές τα κράτη-μέλη Και ε, θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμα. Τελευταία μου ερώτηση. Έχετε την εντύπωση ότι η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω των πολλών μεταναστών που έρχονται στην Ευρώπη. Ήταν καλύτερη θα λέγατε η κατάσταση πριν ε, ξεκινήσει αυτό το κύμα φίξεων. Κατά την προσωπική μου άποψη, όχι. Απλά η κατάσταση γίνεται πιο εμφανή Δηλαδή, εγώ εργάζομαι με τους συνόδευτους ανήλικου εδώ και 15 χρόνια και τα προβλήματα είναι τα ίδια. Πώς θα κρίνουμε την ηλικία, κυδεμόνε, τα ίδια προβλήματα με μικρότερους αριθμού. Και λιγότερα κατά τη μέλη αφορούσε το θέμα ε, του συνήθεις υπόπτου. Το πρόβλημα δεν ήταν τόσο εμφανέ. Οι αριθμοί αυξήθηκαν και αυξήθηκαν γρήγορα, ειδικά σε κάποια κράτη-μέλη. Και πραγματικά έτσι καταλήξαμε στις επιχειρησιακές ε, δυσκολίες. Και Υπάρχουν οι διάφορες ε, δυσκολίες ε, στην εφαρμογή, τι θα ισχύσει, το δίκαιο περί ανηλίκων ή το μεταναστευτικό δίκαιο. Ε, είναι μια μεγάλη πρόκληση. Ακόμα και αν υπάρχει η βούληση και η πόρη, θα χρειαστεί χρόνος. Και σε κάποιες ε, χώρες, αν δούμε το παράδειγμα της Αυστρίας, στην αρχή ήταν μεγάλο πρόβλημα. Ε, παραδείγματος χάρη όλες οι περιπτώσεις ήταν στην Βιέννη η κατάσταση δημιουργήθηκε λόγω της ε, πολιτικής διανομής. Δηλαδή όλες οι περιπτώσεις αυτές ε, μένανε στη Βιέννη. Και μετά πήγαιναν ε, όταν άρχισαν να τα στέλνουν και στα υπόλοιπα κρατήδια υπήρχε κάποια ισορροπία. Κατά την απόψή μου λοιπόν, το πρόβλημα ήταν το ίδιο, αλλά ήταν κρυμμένο. Τώρα, πραγματικά φαίνεται. Και βεβαίως τώρα όλα τα κράτη-μέλη ε, οφείλουν να το αντιμετωπίσουν, δεν μπορούν να το αγνοούν. Και η προλαλή σας έχει δίκιο, το είχαμε αυτό το πρόβλημα. Είχαμε όμως μία περίπτωση ίσως επιτροπίας ε, το χρόνο και λύναμε το πρόβλημα πιο εύκολα. Τώρα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες διαδικασίες ε, και νομίζω ότι τώρα πρέπει να το συζητήσουμε και να το δούμε και να καταλήξουμε κάπου. Και αυτό είναι κάτι θετικό και για τα κράτη-μέλη τα μεμονωμένα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει δηλαδή να αποφασίσουμε κάτι και να το ακολουθήσουμε. Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες αρχές, θα πρέπει να υπάρχει επαφή και με τις ιδιωτικές. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η επικοινωνία τόσο καλή όσο θα έπρεπε. Θα πρέπει να μιλάνε με τους δε. υπάρχει και το πρόβλημα που είναι κάποιοι που δεν είναι μέλη της, της σύμβασης του 1996, υπάρχουν κράτη-μέλη με τα οποία δεν έχουμε συμφωνίες, υπάρχει πρόβλημα με τα έγγραφα που δεν μπορούν να ε, βοηθήσουν, καλό θα ήταν να καταλήξουμε σε μια ομοιόμορφη λύση. Το ίδιο με τις δύο προλαλήσεις, με και εγώ. Έχουν πάρει μεγάλη σημασία λόγω του αριθμού πλέον των υποθέσεων αυτά τα θέματα. Τα κράτη τώρα θέλουν να συνεργαστούν ενώ παλιά το ένα γνώσε το άλλο. Και αυτό οφείλεται στον αριθμό των υποθέσεων. Αλλά είμαστε στην αρχή ακόμα. Ότι είναι ευτυχή συγκυρία ε, μπορεί να φαίνεται λίγο οξύμορο, αλλά πράγματι είναι στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, γιατί τους προσέχουμε ακριβώς χάρη στο μεγάλο αριθμό. Και βλέπουμε την ανάγκη που υπάρχει. Και υπάρχει και προθυμία συνεργασίας πλέον μεταξύ των αρχών που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση και των αρχών που είναι των δικαστικών αρχών που είναι την προστασία των παιδιών. Αυτό είδαμε. Μάλιστα, οπότε μπορούμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Παρά τη δραματική κατάσταση των παιδιών, ε, με θετική νότα. Γιατί ακριβώς αυτό που θέλουμε είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση και κάνουμε αυτές τις προσπάθειες. Σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι και όλες εδώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Να ευχαριστήσω για το θεματικό τμήμα που διοργάνωσε αυτό το εργαστήριο. Πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις και τα briefing paper των ε, κατακλυσμένων μας. Θα τα διαβάσουμε με όλη μεγάλη προσοχή. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα και τους διερμηνείς.